Και αυτό ισχύει για την Ινδία, την Κίνα και άλλες χώρες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σάφη. Ε, βλέπουμε ότι σημειώνεται πρόοδος. Καταδεικνύεται αυτό μέσα στην εκθέση Σας ευχαριστούμε κυρία Ρόιτεβα. Ο συνάδελφος Νικολάσκη.